επιτυχία στο έργο σα. Περισσότερο από ποτέ λέμε έχουμε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, that concludes... Καλώς, έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό που ήταν η ετήσια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή στις 12 σήμερα το μεσημέρι. Στρέφομαι στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία προϋπολογισμού σχετικά με το κοινό σχέδιο λοιπόν, που ενέκρινε η Επιτροπή Συνδιαλλαγής στο πλαίσιο διαδικασίας του προϋπολογισμού 2012 και πρώτο στον κατάλογο μιλητών είναι ο κύριος Λαμασούρ που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ένα λεπτό παρακαλώ. Μπορώ να παρακαλέσω τον κύριο Ντράγκη και τους συναδέλφους τους να συζητήσουν εκτός εθούσης. Ε, είσαστε ευπρόσδεκτος, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε στην εξέταση του επομένου θέματος. Κύριε Λαμασούρα, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως διαπιστώνουμε, η προηγούμενη συζήτηση ε, επηρέασε τα απορέσματα των συζητήσεων του προπολογισμού του 2012 και χαίρομαι γι' αυτό ε, εν τω μεταξύ δεν χαιρετίζουμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου και ε, τον Επίτροπο Λεβαντόσκι και να σας πω τι έγινε σχετικά με τη συνδιαλλαγή για τον προπολογισμό του 2012 που επιτρέπει να κλείσουμε τη διαδικασία στα πλαίσια που προέβλεπε η συνθήκη. Θέλω να χαιρετήσω και να συγχαρώ την Πολωνική Προεδρία που επέ επέτυχε ομοφωνία στο Συμβούλιο και για τον προϋπολογισμό του 2012 και για τον διορθωτικό προϋπολογισμό επαριθμών 6 του 11. Λέγει λοιπόν ότι είναι οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την περίοδο κρίσεως για να συνδυάσουμε δύο αντιφατικούς στόχους οι οποίοι είναι απαραίτητοι. Κατά καταρχήν να μειώσουμε τα έξοδα λειτουργίας και να διατηρήσουμε τα μελλοντικά, τις μελλοντικές δαπάνες για να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα και την αυριανή ανταγωνιστικότητα. Συγχρόνως όμως από αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να συμπεράνουμε τα εξής. Καταρχήν δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε ανάποδα, δηλαδή με ε, ε, ε, πιστώσεις πληρωμών ενώ χρειάζονται πιστώσεις δεσμεύσεων. Πρέπει εμψυχρό τους μελλοντικούς μήλες, μήνες να αξιολογήσουμε την κατανάλωση των πιστώσεων γραμμή προς γραμμή του προϋπολογισμού κατά τρόπο ώστε για τον προϋπολογισμό του 2013 να έχουμε πλήρη ενημέρωση και να μην υπάρχει ενιαίο κούρεμα ή πάγωμα για τρίτη χρονιά. Επίσης δεν μπορούμε πλέον να χρηματοδοτήσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό με εθνικές συνδρομές και από τη Δευτέρα αρχίζουν συζητήσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα ε, νέο τρόπο συλλογής ιδίων πόρων και το επαναλαμβάνω εδώ ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία επί του επομένου δημοσιονομικού πλαισίου χωρίς να επανέλθουμε σε μία πολιτική απόφαση για τη χρηματοδότηση μέσω ιδίων πόρων. Ακούω εδώ πολλούς που θα μιλήσουν για δημοσιονομικό φεντεραλισμό. Όσοι λοιπόν τον εύχονται θα μπορέσουν να τον υλοποιήσουν ευρωπαϊκά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαμασούρ. Για τρία λεπτά έχει το λόγο η κυρία Μπαλσάνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στις 18 Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε μια κοινή θέση για τον προϋπολογισμό λίγες μέρες πριν από το τέλος της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα θα έλεγα σε μια εποχή αβεβαιότητας και δυσκολίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να στραφούν και στο μέλλον τα ευρωπαϊκά όργανα. Είναι επίσης και μια επιλογή ευθύνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ αρχής έθεσε στο κέντρο των συζητήσεων την στρατηγική 2020, την μεγάλη στρατηγική ενάντια στην κρίση για την ευημερία. Δεν είναι εύκολο σήμερα να κάνει κανείς ένα καλό προϋπολογισμό, ούτε καν η Ευρώπη. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε τις επιλογές οι οποίες αναγνωρίστηκαν από όλους κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής. Έχουμε περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη, για την έρευνα, για την εργασία, για τη διαβίου κατάρτιση, για τις πολιτικές μετανάστευσης και για τις διεθνείς πολιτικές. Από τη συνδιαλλαγή βέβαια μερικές φορές τα κοινοβούλια ε, δεν ε, μπορούν να επηρεάσουν όσο θα ήθελαν. Αυτό δεν είναι κάτι το καινοτόμο. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τομέα των πληρωμών, σαν παράδειγμα, ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή από τη μία και το Συμβούλιο από την άλλη. Αυτή η αντιπαράθεση θα πρέπει να ξεπεραστεί γιατί είναι προφανές ότι η κατάσταση που δημιουργήθηκε δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε πλέον στο επίπεδο των πληρωμών. Η ε, συνδιαλλαγή βέβαια δεν είναι και ο καλύτερος πάντα τόπος για να γίνει συζήτηση. Θα πρέπει να υπάρξουν προσπάθειες συμφιλίωσης. Ε, η εμπειρία από πέρυσι μαθαίμαται ότι το να ξεκινούν μεγάλες συζητήσεις μέσα στο χρόνο τον περιορισμένο της συνδιαλλαγής, τον προκαθορισμένο χρόνο, είναι κάτι που επηρεάζει αρνητικά τον προπολογισμό. Οι προβλέψεις για τις ανάγκες της δαπάνες, τις οποίες κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εξαιρετικές προβλέψεις, τις οποίες στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ουσία δεν καλύπτονται. Ελπίζω να βρεθούν κάποιες λύσεις. Μέχρι τη στιγμή κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποκτήσει πραγματικούς ιδίους πόρους, δεν θα λύσουμε αυτό το προφανές πρόβλημα. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα πλαίσια της προσπάθειας την οποία έχουμε αναλάβει δημοσιονομικά, να παρεμβαίνουμε δηλαδή έγκαιρα όταν υπάρχουν ανάγκες σε επίπεδο πληρωμών για την αύξησή τους κατά τη διάρκεια του έτους, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε. Θα πρέπει να τιμήσουμε την υπογραφή μας θα πρέπει να εργαστούμε όλοι έτσι ώστε αυτές οι ανηλυμένες υποχρεώσεις να μην πέσουν θύματα τυπικών διαδικασιών στα πλαίσια της επόμενης δημοσιονομικής διαπραγμάτευσης. Το κάναμε και φέτος με το ίτερ και με άλλες πληρωμές. Θα πρέπει εμείς να αποφύγουμε, να ανοίγουμε συνδιαλλαγές μέσα στην κύρια συνδιαλλαγή. Πάντω, θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου, οι οποίοι με πάθο πήραν μέρο σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία η οποία υπήρξε πρόδρομο στην προσπάθεια έβρεση λύση και τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι ο οποίο κράτησε μια ισόρροπη θέση καθ' όλη τη διάρκεια τη συνδιαλλαγή. Να ευχαριστήσω και τις πολιτικές ομάδες και τους βοηθούς μας οι οποίοι μέχρι τη νύχτα βοήθησαν για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Μπαλζάνη. Το λόγο έχει τώρα για τρία λεπτά ο κύριος Φερνάντες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαιρετίζω εδώ και την παρουσία του Συμβουλίου. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ καταρχήν όλους σας για την δουλειά που έχετε κάνει ετοιμάζοντας τον προπολογισμό αυτό. Χάρη στη δουλειά των πολιτικών ομάδων και των σχεδόν εισηγητών καταφέραμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ για την τόσο καλή συνεργασία που είχαμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου. Υπογραμμίζω επίσης την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε και με το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μα στήριξε επίση η Γραμματεία τη Επιτροπή Προπολογισμών και οι ε, συνεργάτες μας από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και γενικά τις πολιτικές ομάδες. Η δουλειά που κάναμε ήταν ε, μια δουλειά πολύ σοβαρή. Ασχοληθήκαμε με όλους τους τομείς πέρα από τις ε, δαπάνες που απορρέουν από την ένταξη της Κροατίας και την έλευση νέων ευρωβουλευτών. Ασχοληθήκαμε και με υπηρεσίες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και άλλα πράγματα που προβλέπονται από την συνθήκη της Λισαβόνας. Καταφέραμε λοιπόν να καταλήξουμε σε μια αύξηση 1,3%. Παρόλα τα καθήκοντα αυτά τα νέα που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το 2012 ο διοικητικός προϋπολογισμός των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων ε, θα μειωθεί, θα έχει αρνητική αύξηση. Επίσης, χαίρομαι και για τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε την Παρασκευή που μας πέρασε ε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων. Το Συμβούλιο ενέκρινε πλήρω την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τι διοικητικέ δαπάνε και τι λειτουργικέ δαπάνε όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και αναγνώρισε τη λιτότητα και το σωστό της πρότασής μας. Αξίζει τον κόπο αυτό. Ήταν ε, μια δουλειά πολύ σοβαρή που έγινε και που κατάφερε να καταλήξει σε μια ισορροπία ε, μέσω των μειώσεων εκεί που χρειαζόταν, αλλά και της κάλυψης των, δαπαλό, δαπανών εκεί που επίσης χρειάζονται. Όλες οι διοικητικές δαπάνες λοιπόν και οι λειτουργικές όλων των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτω από ένα 6% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 94% ο προϋπολογισμός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για επενδύσεις. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν ανταποκρίνεται σε ένα 1% του ΑΕΠ και αποτελεί μια πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία που προσφέρει μια αλληλεγγύη. Γι' αυτό και πρέπει να ενισχύεται όλος ιδιαίτερος τώρα σε περίοδους κρίσης. Ενισχύονται επίσης οι πιστώσεις για την οικονομική ανάπτυξη, την κατάρτιση, την έρευνα και την νότητα. Θέλω όμως να εκφράσω την ανησυχία μου και να πω στο Συμβούλιο προσοχή. Είναι σημαντικό για την αξιοπιστία μας να φέρουμε σε πέρα στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Οι δαπάνες λοιπόν πρέπει να τηρηθούν έτσι όπως έχουν προβλεφθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους του Συμβουλίου τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ντόμινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, είναι η πρώτη φορά που χρειάστηκε να διαπραγματευτούμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια μιας τόσο σημαντικής ε, κρίσης, σαν και αυτήν την οποία βιώνουμε. Είναι η πρώτη φορά επίσης που νομίζω ότι πετύχαμε μέσα σε συντομότερο ε, χρονικό διάστημα από αυτό το οποίο προβλέπεται στη συνθήκη της Λισαβόνας να καταλήξουμε σε μια πρόταση. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για μια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών οργάνων τα οποία ενεπλάκησαν στη συζήτηση αυτή. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους εγκαρδίους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον πρόεδρο Λαμασούρ φυσικά και την κυρία Μπαλσάνη και τον κύριο Φερνάντες και τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι και τις ομάδες τους. Να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς γιατί πράγματι αντιμετώπισαν το θέμα αυτό με πολύ επικοδομητικό τρόπο. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης του προϋπολογισμού του 2012 ανάμεσά μας ανάμεσα στους αυτούς που πήραν μέρος στις συζητήσεις δεν υπήρξαν πάρα πολύ σημαντικές διαφωνίες σχετικά με το μέλλον του προϋπολογισμού. Υπήρξε μια συζήτηση η οποία ήταν συζήτηση συγκεκριμένη, επαγγελματική θα έλεγα, έτσι ώστε να βρούμε τα μέσα για να κάνουμε πραγματικότητα τον προϋπολογισμό αυτό. Να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας έτσι ώστε η ευρωπαϊκή κοινωνία να νιώσει με τον πιο ευεργετικό τρόπο τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολιτικές να καλύψουν τις ανάγκες εκεί όπου οι ανάγκες είναι οι πιο οξυμένες. Να επιστήσω επίσης την προσοχή σας στο εξής. Προσπαθώντας να απαντήσει κανείς σε αυτό το πνεύμα, να ανταποκριθεί σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας, το Συμβούλιο υιοθέτησε το σύνολο των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των πιστώσεων υποχρεώσεων και ε, των δαπανών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους για την κατανόηση την οποία δείξατε σχετικά και με τις δικές μας προτεραιότητες, τις προτεραιότητες του Συμβουλίου γύρω από τις πιστώσεις πληρωμών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έλεγα ότι τις ανάγκες τις οποίες εκφράσαμε εμείς ε, δεν έγιναν απόλυτα κατανοητές σε σχέση με, ε, τις, ε, με τη σημερινή κρίση. Αλλά παρόλα αυτά υπήρξε μια προσεκτική ανάλυση των προτάσεων του Συμβουλίου. Να σας ενημερώσω επίσης ότι χθε κατά τη διάρκεια του ΕΚΟΦΗΝ το Συμβούλιο υιοθέτησε ομόφωνα τον προϋπολογισμό για το 2012 και με πλειοψηφία υιοθέτησε τον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαρίθμου 6. Λοιπόν, η διαδικασία υιοθέτηση του προϋπολογισμού για το 2012 έχει ολοκληρωθεί με υποδειγματικό τρόπο. Ευχαριστώ ο, κύριος, ε, ο Επίτροπος κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρετίζω τη Συμφωνία για τον Προϋπολογισμό εγκαίρος του Προϋπολογισμού 2012 που είναι ένα ευίωνο σημαδί, μία ένδειξη σταθερότητος στη σημερινή ασταθή Ευρώπη με τόσα ερωτηματικά. Θα ήθελα λοιπόν να πω συγχρόνως και ανοιχτά ότι οι ε, προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της Ευρώπης σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, την ε, ε, πολιτική γυτνιάσεως και επίσης μία επιμονή στην ενίσχυση της Παλαιστίνης. Η έγκαιρη συμφωνία για τον προπολογισμό του 2012 επιτρέπει να εφαρμόσουμε σωστά τον προϋπολογισμό. Και αυτό είναι σημαντικό. Όπως είναι άλλωστε σημαντικό να αυξηθούν τα λειτουργικά, οι λειτουργικές δαπάνες με μία μείωση της ε, ε, διαχειρίσεως. Βλέπουμε ότι υπήρξε μία προσπάθεια να μειωθούν οι ε, οι διαχειριστικές δαπάνες παρόλο που αυξηθήκανε τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσης από 27 σε 28 και πρέπει να χαιρετήσω την ε, επιλογή των ε, προτεραιοτήτων και ε, την έκθεση της κυρίας Μπαλσάνη όπως άλλωστε και τις κινήσεις της διοικήσεως και τον εισηγητή κύριο Φερνάντες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η έγκαιρη συμφωνία δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τον επικοδομητικό ρόλο της Πολωνικής Προεδρίας και του εκπροσώπου της ε, κύριου Ντομινίκ ο οποίος ε, ε, επενεύει <clears throat> στα θέματα του ευρωπαϊκού προπολογισμού σε ορισμένα σημεία το επίπεδο των ε, πληρωμών δεν επαρκεί. Και το επαναλαμβάνω. Και επαναλαμβάνω επίσης ότι εν αντιθέσει με τον ε, ετήσιο προπολογισμό, ανοιχτός προπολογισμό αναφέρεται σε επενδύσεις. Και όταν μιλάμε για επενδύσεις του 2012, στη χώρα που γνωρίζω καλά βλέπω ότι έχουν μειωθεί κατά 5%. 50 ή 60% του ευρωπαϊκού προπολογισμού θα έπρεπε να αποδίδονται μόνο σε επενδύσεις για να καλύψουν το επενδυτικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτρέψουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ε, Αν λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα σήμερα θα το αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον και γιατί και τώρα δεν υπάρχουν ε, επαρκείς πληρωμές και το βλέπουμε στον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 6. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τις πληρωμές και αυτό είναι φυσιολογικό και δεν είναι αξιοπερίεργο. Στην προηγούμενη συζήτηση ένας από τους συζητητές του Κοινοβουλίου είπε στον κύριο Ντράγκη ότι πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ πιστεύω ότι έγινε μία δήλωση ότι αν χρειαστούμε άλλα χρήματα για το 2012 θα ευρεθούν και θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλες τις προσωπικότητες οι οποίες ενεπλάκησαν όπως ο κύριος Λαμασούρ και επέτυχαν τη συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2012. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Περνάμε στους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Πρώτα, ο κύριος Λαβία, εκ μέρους του Αλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να μου επιτρέψετε εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο να ευχαριστήσω του εισηγητές Μπαλζάνη και Φερνάντε, και τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι. Όπω και τον Πρόεδρο Ντομινίκ, τον, πρόεδρο, τον εκπρόσωπο της Προεδρίας του Συμβουλίου, τον κ. Ντομινίκ, για το πνεύμα συνεργασίας κυρίως, το οποίο επέδειξαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η συμφωνία της παρασκευή 18 του μηνό το βράδυ είναι μια καλή συμφωνία, είναι ένα καλό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την τρομερή κρίση την οποία αντιμετωπίζουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Σε σχέση με τις πιστώσεις υποχρεώσεων είμαι ικανοποιημένος από την απόφαση που ελήφθη για να χρησιμοποιηθεί το μέσο ευελιξίας για 200 εκατομμύρια στον τίτλο 4, όπως το είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάκαμψη του παραγωγικού συστήματος, για τη χρηματοδότηση των κατά προτεραιότητα καθορισμένων πολιτικών, σεβόμενη το κέντρο, τον πυρήνα της στρατηγικής του 2020 και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που θέτει η πολιτική γειτονία. Είναι επίσης σαφές ότι οι υπόλοιπε πολιτικές σε επίπεδο υποχρεώσεων βλέπουν τις ανάγκες τους να καλύπτονται από τις προτεραιότητες τις οποίες θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές όμως ότι οι πιστώσεις πληρωμών, όπως το είπαν και πάρα πολλοί συνάδελφοι κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συζητήσεων και από τους ίδιους τους εισηγητές, δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικοί. Ιδιαίτερα σε σχέση με την διαφορά η οποία αυξάνεται ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις πληρωμές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας δημιουργήσει δυσκολίες. Θα δημιουργήσει δυσκολίες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποια από τα προγράμματα τα οποία προχωρούν. Πιστεύω λοιπόν ότι η ψηφοφορία σήμερα στο Κοινοβούλιο όπως και η χθεσινή ψηφοφορία στο Συμβούλιο θα καταστήσει τον προϋπολογισμό μας αποτελεσματικό, θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την κρίση, θα επιτρέψει την ανάκαμψη των επενδύσεων στην οικονομία για μια έξυπνη και διαρκή ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λαβία. Το λόγο τώρα εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχει για δύο λεπτά ο κύριος Φάρμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την Πολωνική Προεδρία όπως επίσης και τους εισηγητές μας, Μπαλτσάντη και Φερνάντες. Μετά από μια μακρά διαπραγμάτευση καταλήξαμε σε συμφωνία και τη στηρίζω τη συμφωνία αυτή, γιατί καταφέραμε να πετύχουμε πολλά για την κατάρτιση, για τις πολιτικές γυτνίασεις κλπ. Μπορώ να υποστηρίξω λοιπόν τη συμφωνία αυτή. Οι διαπραγματεύσεις όμως οδήγησαν και στην αποκάλυψη θα έλεγα πολλών ανησυχιών για το μέλλον και πολλές διαφορές φάνηκαν στο εσωτερικό, μάλλον και πολλές απόψεις διαφορετικές ακούστηκαν και στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων και της ομάδας της Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής Ομάδας. Ξέρω ότι πάρα πολλές χώρες, όπως η δική μου, ιδιαίτερα οι χώρες οι οποίες συνεισφέρουν θετικά στον προϋπολογισμό, δεν βοηθούν για να υπάρξει μια σωστή πολιτική που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα στο μέλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο προπολογισμό αν πράγματι θέλουμε να ανακάμψουμε, αν πράγματι θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση στι χώρε οι οποίε το χρειάζονται περισσότερο. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε καλύτερα λοιπόν αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί. Πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μα στην εφαρμογή, στι πληρωμέ και να καλύψουμε σωστά τα χρέη μας μέσα σε ένα έφετο χρονικό διάστημα. Κάποιες χώρες όμως όπως είπα έχουν μια αρνητική αντίληψη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα μας επηρεάσει πάρα πολύ άσχημα στο μέλλον. Κάποια κράτη-μέλη θα προσπαθήσουν να παγώσουν ας πούμε τον τη συμμετοχή τους στον προϋπολογισμό στη Γεωργία να μην υπάρξουν νέοι πόροι για έναν τομέα ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, οι υποδομές, οι έρευνες για το κλίμα και τις κλιματολογικές συνέπειες των αλλαγών. Λοιπόν, είναι σαφές ότι μια πλειοψηφία βέβαια στο Κοινοβούλιο και μια πλειοψηφία κρατών μελών μπορούν να συμφωνήσουν σε θετικά μέτρα. Ελπίζω η Πολωνική Προεδρία και η επερχόμενη Προεδρία της Δανίας να ξεπεράσουν αυτήν την μειοψηφία η οποία μπλοκάρει την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριος Χάκλοντ από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από οτιδήποτε άλλο θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές της ομάδας του Κοινοβουλίου. Η πολιτική μας ομάδα, οι φιλελεύθεροι, θα υποστηρίξουν την συμφωνία η οποία θα τεθεί προς ψηφοφορία αργότερα σήμερα. Ε, ε όταν εξετάζαμε το θέμα της διαπραγματευτικής εντολής, είχαμε δει ότι υπήρχε πιθανότητα μερικές φορές να απορρίψουμε την πρόταση του προϋπολογισμού τα πράγματα άλλαξαν κάπως και είναι προφανές βέβαια ότι ένα 5% αύξηση ε, δεν θα μπορούσε να γίνει εύκολα δεκτό κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Αλλά αυτό το 2 και κάτι της 100 νομίζω ότι είναι πιο κατανοητό και μπορεί να γίνει γενικότερα δεκτό σήμερα. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φάρμ για την διαβίου κατάρτιση, για την έρευνα και την ανάπτυξη είναι σωστά. Ταυτόχρονα, όπως και στους τομείς των πολιτικών εξωτερικής πολιτικής, ε, βλέποντας το τι γίνεται στη Βόρεια Αφρική σαν παράδειγμα, βλέποντας το τι πρέπει να κάνουμε και εμείς σε σχέση με τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, θα δούμε ότι όλα αυτά έχουν οικονομικές συνέπειες. Εν πάση περιπτώσει είναι καλό το ότι ψηφίστηκε, φτάσαμε ως εδώ στα πλαίσια του προϋπολογισμού σήμερα. Πρέπει να δούμε όμως τι θα γίνει στο μέλλον. Ακούσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα στο Συμβούλιο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διστάζουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει και αυτό μας ανησυχεί επαναλαμβάνω για το μέλλον. Φυσικά και έχουμε μια κάποια συμφωνία για τον προϋπολογισμό. Ήταν απαραίτητο να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία κατά από τις παρούσες συνθήκες. Αλλά λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στο Συμβούλιο θα δούμε ότι στο μέλλον κάτι τέτοιο να μην είναι τόσο εύκολο αν θέλετε. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσει και το Συμβούλιο ποια είναι η πραγματικότητα και να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ κύριε Χάκλον. Για τους Ευρωπαίους μεταρρυθμιστές συντηρητικούς, ο κύριος Βανόρτεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, το Κοινοβούλιο δέχτηκε ε, μία αύξηση η οποία είναι χαμηλότερα από το 2011 αλλά έχασε και την ευκαιρία να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Δηλαδή ε, είναι σαν να λέμε ότι είχαν χρησιμοποιηθεί σωστά στο παρελθόν οι πόροι ενώ βλέπουμε ότι τα κράτη μειώνουν τους προϋπολογισμούς για να μειώσουν τα ελλείμματα και δεν μπορούν να προκαλέσουν ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά η όρεξη των χωρών αυξάνεται και έπρεπε να υπάρξει σημαντική περικοπή του κοινοτικού προϋπολογισμού να επιστραφούν πόροι ή στα ταμεία των κρατών ιδίως για τους τομείς ερεύνης και αναπτύξεως. Ενώ διαμέσου των των αυξάνονται οι αρμοδιότητες σε που δεν θα χρειαζόταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προβεί σε σημαντικές περικοπές και ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι ένα μικρό ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού αλλά ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια το χρόνο που θα μπορούσαμε να έχουμε περικόψει περίπου το 1 τέταρτο και ε, να έχουμε ε, περιορίσει σημαντικά χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία. Ε, συντηρούμε την γραφειοκρατία του Κοινοβουλίου διότι αντιλαμβάνουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει ε, ή νοικιάζει κάπου 62 κτίρια δεν υπάρχει καμία περικοπή και έχει φτάσει η ώρα να προβούμε σε μεγαλύτερη λιτότητα. Ευχαριστώ η κυρία Τρίπελ τώρα για 4,5 λεπτά εν ονόματι των Πρασίνων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός για το 2012 σημερινή έναν προϋπολογισμό εξοικονόμησης και το πολιτικό ερώτημα που θέτουμε και πρέπει να απαντήσουμε είναι αν είναι ένας σωστός προϋπολογισμός ο οποίος είναι φιλικός προς το περιβάλλον, και της Ευρώπης διότι ε, πρέπει να καταρτήσουμε νέες προτεραιότητες δεν πρέπει να μειώσουμε τις βιώσιμες πολιτικές ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτε στη γεωργία ούτε στη, στα διαρθρωτικά ταμεία αλλά να, μη, να αναπτύξουμε ε, ανταγωνιστικές πολιτικές διότι ακούσαμε ε, ότι το 2000 10 αυξήθηκαν ε, οι εκπομπές διεξιδίου του άνθρακος διεθνώς κατά 6%. Δεν θα μπορέσουμε έτσι να προστατεύσουμε τον πλανήτη. Και ε, ακόμη και στο θέμα αυτό δεν ε, προσφέρουμε επαρκή. Και θα έπρεπε να σας πω ότι εγώ έρχομαι από το μικρότερο κρατήδιο της Γερμανίας τη Βρέμη και εδώ και χρόνια εφαρμόζουμε μία πολιτική και ξέρω γιατί μιλώ. Δεν είμαι από άλλο πλανήτη, ξέρω τι γίνεται, αλλά οι προπολογισμοί των τελευταίων των διαφόρων κρατών μελών τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε και υπάρχουν λόγοι να πούμε ότι όντως ε, ορθά ο μικρότερος προϋπολογισμός ε, ε, αντιπροσωπεύει 1% και πρέπει να αυξήσουμε παραδείγματος χάρη ε, τις προοπτικές του μέλλοντος που δεν υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέρη και εκεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να επηρεάσει θετικά αλλά έχουμε 25 εκατομμύρια για τις νέες εποπτικές αρχές για να ρυθμιστούν καλύτερα οι Υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα για τις ψηφιακές αγορές και στο διοικητικό προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου υπήρξε ε, μια ε, περικοπή στις ε, δαπάνες διερμηνίας και μετάφρασης και ταξιδίων. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στον περιορισμό και δίνουμε έτσι το σήμα προς τον Ευρωπαίο πολίτη και στη δημοσιότητα. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω ιδίω τους εκπροσώπους του Συμβουλίου ο προϋπολογισμός αυτός εξασφαλίζει ε, τις ε, βιώσιμες προοπτικές της Ευρώπης διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ε, την διάσκεψη στον Τέρμπαν, το είπε και ο κύριος Λεβαντόσκι πρέπει να υπάρξει ένας επενδυτικός προϋπολογισμός που να χρησιμοποιηθεί σωστά να υπάρξουν νέα κίνητρα για νέα βιώσιμα προϊόντα για νέες, για τεχνολογίες βιώσιμες, για νέα προϊόντα, διότι μόνο έτσι θα προχωρέσει η Ευρώπη και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία και μία τέτοια πορεία δεν την ε, διαπιστώνω στον προϋπολογισμό. Πάντοτε λοιπόν μας λέγατε εξοικονομήστε, εξοικονομήστε και όταν αναφερόμαστε στον αντιδραστήρα χάσεως ο οποίος ενδέχεται κάποτε να λειτουργήσει ε, θα ε, δαπανίσουμε 1,3 περισσότερα δις για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι λογικό, δεν θα έπρεπε στο μέλλον να ε, εξετάσουμε περισσότερο την, στην έρευνα τομής που ξέρουμε ότι θα επιτύχουμε αντί αυτών τον αντιδραστήρα που δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε Επίση, επίσης υπάρχει η δήλωση ε, του Συμβουλίου ότι θα πρέπει ε, να υπάρξει χρηματοδότηση η οποία δεν είναι σαφής και γι' αυτό η πολιτική μου ομάδα δεν είναι σε θέση να ε, υπερψηφίσει αυτόν τον προϋπολογισμό. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ανατολικής Αριστεράς και Συμμαχίας των Βορείων Χωρών για 1,5 λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Πόρτας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά, το 2012, δεν θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Για την έρευνα, κύριε Λεβαντόφσκι, για την οικολογία, για την κοινωνική αλληλεγγύη, ο προϋπολογισμός αυτός, τα κεφάλαια αυτά, δεν είναι αρκετά δυνατός. Ούτε διορθώνει τις εθνικές πολιτικές, ούτε τις βοηθάει που είναι πολιτικέ λιτότητας και συνεχίζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα προπολογισμό ο οποίο δεν αναγνωρίζει την ύφεση στην Ευρώπη. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία, την φτώχεια, ιδίω μεταξύ των νέων. 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ δίνουμε, λιγότερο δηλαδή από ό,τι στον προπολογισμό του 2011. Ένα ελάχιστο δηλαδή για μια ελάχιστη Ευρώπη. Κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Business as usual. Πρόεδρε, θέλουμε να αυξήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις πληρωμές, από ό,τι φαίνεται. Είναι ένας προπολογισμό με κακή δημοσιονομική πρακτική. Θα έπρεπε με μεγαλύτερη σαφήνεια να είχαμε καθορίσει τις προτεραιότητές μας στις ε, επενδύσεις. Με τον προπολογισμό αυτό ε, θα έπρεπε να, ε, μάλλον αυξάνονται οι πιστώσεις για στρατιωτικές έρευνες, για την Frontex. Στηρίζουμε τις εξαγωγές που καταστρέφουν τις υπονάπτυξη χώρες. Πρόεδρε, και θα τελειώσω με αυτό. Πρόκειται για μια σχιζοφρένεια η οποία υπερισχύει. Όλοι λέμε ότι θέλουμε μια καλύτερη Ευρώπη, αλλά τελικά το επιδόρπιο είναι λιγότερη Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Από το EFD για ένα λεπτό η κυρία Αντρέας, αν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ζήτησαν 5% αύξηση για το 2012. Γελίο. Η αποδοχή από πλευρά του Συμβουλίου ε, για 2% αύξηση είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο των φορολογουμένων Ευρωπαίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ουσία έχει εξοδέψει στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας τρία δις, επαναλαμβάνω. Ένα μάλλον ε, τρεις έχει εξοδέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έχει χάσει τα χρήματα αυτά και ζητάει όλο και περισσότερα. Η σημερινή οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη αντικατοπτρίζει, θα έλεγα, ε, μια φρικτή αποτυχία. Εφόσον αυτές οι δαπάνες οι αδικαιολόγητες συνεχίζονται, ο κύριος Όσμπορν στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώνει ακόμα περισσότερες ε, περικοπές. Όχι κύριε Χέγκ, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν τον ελέγχεται. Κύριε Κάμερον, μια αύξηση 2% δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Επιτέλους, σταματήστε να στέλνετε τα χρήματα των Βρετανών φορολογούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Εκ των μη γεγραμμένων για 1,5 λεπτό, κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ. Το 2012 παρόλες τις, τις κριτικές είναι ένας προϋπολογισμός περικοπών που αποδεικνύει στους πολίτες ότι στις δύσκολες εποχές το Κοινοβούλιο ξέρει να ρυθμίζει τα οικονομικά του διότι 24% του προπολογισμού ωραίουν προς τους πολίτες. Ένα ποσοστό αναφέρεται στα θεσμικά όργανα και επιπλέον για το 2012 έχουμε ε, ένα 8% πράγμα το οποίο ε, αποκρίνεται στις επιθυμίες των κρατών μελών. Να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα μέλλον μετά την κρίση. Ε, ε, έχουμε μεγάλη ανεργία των νέων, ιδίως για τις επόμενες γενιές. Αυτό θα φέρει προβλήματα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο ισχυρή από πλευράς εκπαιδεύσεως και να επενδύουμε για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα παραδείγματο χάρη έχει πολλές δυνατότητες. Ας επενδύσουμε εκεί σε ηλιακή ενέργεια που θα δημιουργήσουμε όχι μόνο βιώσιμες θέσεις εργασίας αλλά και μία πρόοδο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων και τέλος θέλω να ευχαριστήσω ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές και όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βέρτμαν. Περνάμε στους άλλους ομιλητές. Ο κύριος Γαρίγα έχει πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Η άσκηση αυτή ήταν ε, δύσκολη τόσο για την κυρία Μπασάντη όσο και για τον κύριο Φερνάντε. Δύσκολη δουλειά και για την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνδιαλλαγή με επικεφαλής τον κύριο Λαμασούρ. Η Προεδρία του Συμβουλίου φαντάζομαι ότι θα είναι ικανοποιημένη και έχει λόγους γιατί ε, προστάτευσε το δικό της match ball στο αγώνα τένις που είχαμε την βραδιά της συνδιαλλαγής με τον διορθωτικό προπολογισμό αριθμό 6 και τις οικονομικές επιπτώσεις του σχεδίου ΙΤΕΡ. Όμως δεν βλέπω άλλους λόγους για ικανοποίηση. Άλλαξαν για δεύτερη φορά οι κανόνες, οι μη γραπτοί κανόνες της διαπραγμάτευσης για τον προπολογισμό. Πριν αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας, στην συνδιαλλαγή για τον προπολογισμό καθορίζαμε ένα επίπεδο πιστώσεων δεσμεύσεων και μετά αποφασίζαμε για τις απαραίτητες πληρωμές. Τώρα το Συμβούλιο μονομερός βάζει το επίπεδο των πληρωμών και μετά διαπραγματεύεται για τις πιστώσεις. Και για να γίνει αυτό σημαίνει ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπαίνει προ τετελεσμένου γεγονότος. Αυτή τη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δέχεται επειδή βρισκόμαστε σε μια έκτακτη οικονομική κατάσταση επειδή είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία, ακόμα και αν αυτή είναι μια κακή συμφωνία. Όμω αυτό ο τρόπο διαπραγμάτευση, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τίποτα καλό δεν προαναγγέλει για τι επόμενε ε, διαπραγματεύσεις που θα είναι για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά το λόγο έχει τώρα ο κύριος Βόαν. Ε, ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, έτσι και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συγητές για την τόσο καλή δουλειά που έκαναν για την εκπόνηση του προπολογισμού αυτού. Αλλά θέλω να πω δύο λόγια πρώτα απ' όλα για το γενικό προπολογισμό και μετά θα μπω στο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά λοιπόν τον γενικό προπολογισμό, θα έλεγα ότι στηρίζω την συμφωνία στην οποία καταλήξαμε στη συνδιαλλαγή, αλλά έχω και κάποιες ανησυχίες. Ιδιαίτερα με απασχολεί το θέμα ότι στην συνδιαλλαγή συμφωνήσαμε για έναν προπολογισμό ο οποίος δεν δίνει αρκετά χρήματα στα διαφορετικά ταμεία στο μέλλον και τώρα θα έχει και επιπτώσει στι περιφέρειες και σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είναι η Ουαλία για παράδειγμα. Στην Ουαλία εποφελούμεθα κατά πολύ από τα διεθνωτικά ταμεία. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για τα διεθνωτικά ταμεία το 2012 θα φταίει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να καταλάβει και να αναγνωρίσει ότι τα ιδιωτικά ταμεία αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι το Συμβούλιο φταίει. Τώρα για τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι δικιά μου κυρίω ευθύνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι έκανε τη δικιά του τη δουλειά για τον προπολογισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε για ένα μεγάλο ποσοστό ε, περικοπές. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσης δέχτηκαν οικονομίες. Δέχτηκαν πάγωμα των αποζημιώσεων τους για τα γραφεία τους, για τα έξοδα μετακίνησης κλπ. Το κάναμε αυτό. Οπότε για μένα, Πρόεδρε, το σημαντικό μήνυμα του προπολογισμού αυτού είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τις προτεραιότητές του. Αναγνωρίζουμε ότι η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι λεφτά στην απασχόληση και την ανάπτυξη και συγχρόνω οικονομίες εκεί όπου μπορούν να γίνουν πραγματικά οικονομίες. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Άλβαρο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητέ οι οποίοι ε, μαζί με τον κύριο Λαμασούρ έκαναν τόσο καλή εργασία. 17 ώρες χρειαστήκαν οι δύο αυτές ε, ερευνητικέ ε, διαδικασίες και από τις οποίες ήταν δύο ώρες συζητήσεων με το Συμβούλιο. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διαδικασία διαβούλευσης για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Αυτό διευκολύνει τη θέση όλων μας. Παρά το γεγονός ότι καθυστερήσαμε λιγάκι την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε συμφωνήσει όλοι, έχουμε προσεγγίσει τη θέση του, κοινο, του του Συμβουλίου για τις, ε, πληρω... για τις πιστώσεις πληρωμών που περιορίζεται η αύξησή του σε 2,9 δισεκατομμύρια μονάχα και δεχτήκαμε από κοινού με το Συμβούλιο και ένα κοινό επίπεδο για τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Επομένως έχουμε αποφύγει μια σύγκρουση, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν θα τα αποφύγουμε. Δεν μπορεί το Συμβούλιο να συνεχίσει να χρηματοδοτεί με διορθωτικούς και συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς. Υπάρχουν τομείς οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώνονται πάντα με διορθωτικούς προϋπολογισμούς γιατί έτσι σπρώχνουμε το πρόβλημα μονάχα μπροστά μας στο μέλλον. Θα πρέπει κάποτε να ενταχθούν και στον πραγματικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει όλοι ότι χρειάζεται περισσότερα κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη και πρέπει να υποστηριχθεί σε αυτά και από τα κράτη-μέλη. Δεν έχει νόημα να υπάρχει ε, συζήτηση για τον προπολογισμό όταν εμείς <clears throat> είμαστε κλειδωμένοι σε μια λογική μονάχα επιδότησης και δεν θέλουμε να επιτύχουμε συγκεκριμένους στόχους. Με τη λογική αυτή δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιτύχουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020. Είναι απαραίτητο επίσης οι πολίτες να καταλάβουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους υποστηρίζει στην προσπάθειά τους να υπάρξει μια έξοδος από την κρίση και μια ανάπτυξη. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φερνάντες. Έχουμε καταλήξει σε ένα καλό αποτέλεσμα ψηφίζουμε τώρα θετικά για αυτή τη στάση, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να επανέλθουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Άλβαρο. Δίνω το λόγο τώρα για ένα λεπτό στον κύριο Βλάσακ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. υπήρξε μια συμφωνία για τον προπολογισμό του 2012, αλλά αυτό δεν ήταν εύκολο εγχείρημα. Ξέρουμε ότι με μια πολύ μικρή πλειοψηφία μονάχα ενεκρίθη αυτό ο προπολογισμό. Οι πιστώσει πληρωμών είναι λίγο περισσότερο από τα 129 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,6% μονάχα και αυτό καταδεικνύει τις προσπάθειες εδραίωσης των προϋπολογισμών σε εθνικό επίπεδο και την ζωφερή κατάσταση την οικονομική στην οποία βρισκόμαστε σήμερα στην Ευρώπη. Για να τα θέσω τα πράγματα με απλό τρόπο οι πιστώσει πληρωμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε αυτή την κρίση μένουν σε χαμηλό επίπεδο, κάτω από το επίπεδο του προπολογισμού ω αύξηση. Για μένα, ο συντονιστή τη ομάδα μου στην Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων, αυτό εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα, γιατί όταν θέλουμε να πετύχουμε να ακολουθήσουμε τους στόχους μας θα πρέπει για το 2012 να έχουμε αρκετά ποσά για τον τομέα 1β, τον τομέα συνοχής, ώστε με τον τρόπο αυτό να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις πολιτικές μας και να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας από τα προηγούμενα χρόνια. Η κύρια προτεραιότητά μας είναι η κοινή δήλωση για τις πληρωμές στο σημείο 3.1 που που θα εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βλάσακ. Για ένα λεπτό ο κύριος Φιρέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο μας έφερε αποτελέσματα τα οποία μπορούσε κανείς να περιμένει. Έγινε αυτή η γνωστή ιεροτελεστία όπου οι λεγόμενοι ευρω... ευρωπαϊστές τύπτουν το στήθος τους για ένα ισχυρό προϋπολογισμό για μεγάλη αύξηση των κονδυλίων αλλά τελικά καταλήγουν χωρίς καμιά ντροπή να ψηφίζουν την πρόταση του Συμβουλίου, που σημαίνει μια αύξηση μονάχα κατά 1% του προϋπολογισμού και σημαίνει ότι δεν φτάνουμε καν το επίπεδο του, του πληθωρισμού. Ενώ συγχρόνως έχουμε να κάνουμε με τα στραγγαλιστικά εργαλεία, όπως είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο μειώνει στα κράτη-μέλη σε σχεδόν στο μηδέν το, την αναδιανεμητική λειτουργία του προϋπολογισμού που θα ήταν απαραίτητη για να μπορέσουν να μειωθούν οι ανισομέρειε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πολύ καλό, κακό μήνυμα για τι χώρε, οι οποίε είναι τα θύματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των συστημάτων λιτότητας. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ψέμα η λειτουργία του προϋπολογισμού. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ψέμα το οποίο θα διωγγώσει ακόμα περισσότερο τις διαμαρτυρίες στους δρόμους της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει τώρα ο κύριος Χάρτογκ. Πρόεδρε. Ένα Κινέζος επενδυτή πριν από δύο εβδομάδες είπε το εξή. Τα προβλήματα που συνεχίζονται στις ευρωπαϊκές χώρες απορρέουν από μια κοινωνία που είναι σε αδιέξοδο και ζει από σοσιαλιστικές κατακτήσεις. Αντί να εργάζονται, παραμένουν οκνηροί και το σύστημα έχει εκτροχιαστεί. Είναι σοσιαλιστικής προέλευση και έμπνευση και ο προπολογισμό του 2012 και νέε πατάλες και νέε δαπάνες. Η σοσιαλδημοκρατία ε, προσπαθεί να υπερπροστατεύει τα ίδια τη τα συμφέροντα και καταστρέφει ε, την κατάσταση και το βλέπουμε και το 2012 στον προπολογισμό. Αυξάνεται και πάλι ο προπολογισμό και ε, δίνει περισσότερε θέσει απασχόληση στην Ευρωκλίκα που έχει σημαδεμένη την τράπουλα ο προπολογισμό του 2012 δεν είναι προστιθέμενη αξία, δεν οδηγεί στη λύση των προβλημάτων αλλά στην επιδείνωσή τους. Η μόνη λύση που χρειάζεται η Ευρώπη είναι εξοικονόμηση σε άχρηστα πράγματα για να τονωθεί η απασχόληση και να μπορεί ο Κοσμάκης να εργάζεται και να βγάζει τίμια το ψωμί του για να ζει την οικογένειά του. Όλα αυτά δεν γίνονται με τον προϋπολογισμό του 2012. Κάνετε λάθος και εργάζεστε για την καταστροφή της Ευρώπης. Δεν το επιθυμεί αυτό το κόμμα μου, το ΠΒΒ, το κόμμα της Ελευθερία και τη Δημοκρατίας. Γι' αυτό εξ ονόματο των ε, Ολλανδών πολιτών θα καταψηφίσουμε αυτό το προπολογισμό. Ευχαριστώ κύριε Χάρτον. Για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Σούριαν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Τα πρώτα καλά νέα είναι ότι επιτέλους επετέφθη συμφωνία μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και μπορεί επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση του χρόνου να λειτουργεί σωστά. Ως Ούγγρος θα μπορούσα ίσως να προσθέσω ότι οι πιο σημαντικές γραμμές του προπολογισμού κατά την άποψή μας παρέμειναν άθικτες από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή γεωργική πολιτική, η οποία θα συνεχιστεί ως έχει, τα κονδύλια για τη σύγκληση αυξήθηκαν κατά 9%. Τώρα μπορεί κανείς να το συζητήσει αυτό, είναι πολύ λίγο. Αλλά νομίζω ότι ευθυγραμμίζεται με την πραγματικότητα. Υπάρχουν και κάποια άλλα μικρότερα στοιχεία που μπορεί να μας χαροποιήσουν, όπως είναι η αύξηση κατά 9 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος παροχής γάλακτος στο σχολείο. Πάντως, και σε κάποια άλλα δεν έχουν αυξηθεί οι πιστώσεις, για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγκρίναμε ένα πρόγραμμα στον τίτλο για τον πολιτισμό για να ε, σωθούν μειονοτικές γλώσσες και λιγότερο μιλούμενες ε, γλώσσες που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις λύσεις που θέλουμε να εφαρμόσουμε και να τερματιστεί η κρίση. Λοιπόν, αν κανείς σταθμίσει την κατάσταση, βάλουμε από τη μία τα θετικά του προπολογισμού και από την άλλη τα αρνητικά και τα συγκρίνουμε, θα έλεγα σε τελική ανάλυση ότι το ποτήρι είναι 80% γεμάτο και 20% άδειο. Χρειάζεται λίγη δουλειά ακόμα για να το γεμίσουμε μέχρι πάνω, αλλά αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα φυσικά και θα υποστηρίξει τον προπολογισμό. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει τώρα η κυρία Γκαρδιά Σάμπαλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε πολλές λεπτομέρειες και ίσως με τον τρόπο αυτό χάνουμε το δάσος για τα δέντρα. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν επικρίνει το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων, αλλά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να τονιστεί, θα μπορούσε να τονιστεί ότι συνέπιπταν κατά 95%. Αν δούμε λοιπόν την ε, τη διαδικασία αυτή σε σχέση με τα τελικά αποτελέσματα δεν ήταν κακό το αποτέλεσμα. Έχουμε περάσει προγράμματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την κρίση για το επιχειρήν και την καινοτομία, για την ευφυά ενέργεια, προγράμματα όπως το Erasmus Mundus. Και επίσης έχουμε εξασφαλίσει και χρήματα για να βοηθήσουμε τους ε, γείτονές μας από την νότια όχθη της Μεσογείου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα μέλλον πιο δημοκρατικό. Το Συμβούλιο εδώ και τρία χρόνια λέει μονάχα ένα πράγμα. Λιτότητα. Και δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να αλλάξει γνώμη. Αν λοιπόν δεν υπήρχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε δεν θα μπορούσαμε να αναχαιτήσουμε τα αποτελέσματα τα οποία βλέπει η Ευρωπαϊκή Ήπειρος σε επίπεδο εθνικών κρατών λόγω της λιτότητας. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα βήμα ακόμα προς τα εμπρός. Ένα πράγμα είναι το να μειώσουμε τις πιστώσεις πληρωμών και το άλλο είναι να μην τηρήσουμε τις υποχρεώσεις οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή ε, συναυθεί και πρέπει να εκπληρωθούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήνουμε τις υποσχέσεις μας και να μην τις πραγματοποιούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκάρδια αλλά Η κυρία Γένσεν για δύο λεπτά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου σε σχέση με τα αποτελέσματα τα οποία επιτέθησαν στη διαδικασία του προϋπολογισμού. Το Κοινοβούλιο πιστεύω ότι κατάφερε να εξεύρει κονδύλια για την χρηματοδότηση της ε, Παλαιστίνης, να βρει τα απαραίτητα κονδύλια για το ΙΤΕΡ, για την θερμοποιηνική σύνδεξη, χωρίς να θίξει παρόλα αυτά το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Παρ' όλα αυτά, εγώ νιώθω κάποιε ανησυχίε για τον διορθωτικό και συμπληρωματικό προπολογισμό υπαριθμών 6. Νομίζω ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε δεν είναι πια κάτι το οποίο μπορούμε να αντέξουμε. Από τη μια μεριά, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη λένε ότι αν χρειαστούμε συμπληρωματικό προπολογισμό θα τον ε, εγκρίνουμε. Και η Κομισιόν από την άλλη πλευρά μας τονίζει ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα χρήματα για να πληρώσουμε αυτούς τους λογαριασμούς και μας λένε τα κράτη-μέλη, όχι, όχι, δεν είναι σωστή η λογαριασμή της Κομισιόν, δεν χρειαζόμαστε τόσα λεφτά και δεν λένε συγχρόνως τι θα ήταν τα σωστά αριθμητικά στοιχεία. Αυτό είναι μια απαράδεκτη κατάσταση, μια αφόρητη κατάσταση. Όταν λοιπόν κανείς αναλαμβάνει κάποιες υποχρεώσεις θα πρέπει να τις στηρίζει ως το τέλος. ο προϋπολογισμός που έχουμε ενώπιόν μας είναι ένας προϋπολογισμός υποχρεώσεων κατά που έχει μελλοντικές επενδύσεις. Δεν έχει άμεσες πληρωμές αυτή τη στιγμή, αλλά οι πληρωμές αυτές θα έρθουν εν καιρό. Εγώ πήρα μετά από την έγκριση του προπολογισμού ένα email από ένα δανεικό κέντρο έρευνας που μου εξηγούν ότι είναι όλο και περισσότερο δύσκολο να πάρουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθυστερούν όλο και περισσότερο οι πληρωμές. Βλέπω λοιπόν ότι εδώ αρχίσουμε να σπρώχνουμε μπροστά μας τις δύσκολες αποφάσεις και να τις αναβάλουμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπομισθούμε τις ευθύνες μας και να πληρώσουμε τη νύφη. Η κυρία για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται θετικά νέα και καλές ειδήσει αυτό τον καιρό. Και το γεγονός ότι τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν για τον προπολογισμό του 2012 είναι καλά νέα. Θα ήθελα λοιπόν επ' να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν για το έργο τους και ιδιαίτερα τους συνεργάτες μας, τους βοηθούς μας, ε, τους υπαλλήλους της γραμματείας που πολύ συχνά ξενύχτησαν Μέχρι τις μικρές πρωινές ώρες ε, εργάζομαι. Δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι τα σημαντικότερα δημοσιονομικά προβλήματα βεβαίως δεν έχουν λυθεί. Επιπλέον, βλέπουμε καλύτερα ε, ορισμένα προβλήματα που πρέπει να λυθούν όταν συζητούμε για τον προπολογισμό και ελπίζω να λυθούν το συντομότερο. Παράδειγμα, ο διορθωτικός προπολογισμός υπαριθμών 6 για το 2012. Χαίρομαι που βρήκαμε μια συμφωνία και γι' αυτόν, αλλά ο τροποποιητικός αυτός διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 6 κατέδειξε ορισμένα προβλήματα, τα οποία συνειδητοποιήσαμε, τα οποία θα παραμείνουν και μάλιστα θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερα σε σχέση με τα όσα σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα κοινό διπλωματικό σώμα, ας πούμε, ή ε, ζητήματα ανθρωπιστικής βοήθειας, διαφορετικές ε, μεταρρυθμίσεις, έρευνα και ανάπτυξη. Θα μπορούσα να συνεχίσω να παραθέτω ακόμα πολλά θέματα. Δυστυχώς, για όλες αυτές τις προσδοκίες... Δεν ε, έχουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί συνεχώ σε νέε δράσει χωρί να προσθέτει και του απαραίτητου οικονομικού πόρου. Ελπίζω κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να συνεχιστεί ο διάλογος και για τις πληρωμές, για τα θέματα που σας ανέφερε. Και με χαρά θα συμμετέχω στο διάλογο αυτό. Σα ευχαριστώ και πάλι και ελπίζω η συνδιαλλαγή να προχωρήσει. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό, κυρία Γκρελιέ, έχει το λόγο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό ο προπολογισμό 2012 είναι τελικά ο προπολογισμό του Συμβουλίου, στο οποίο το Ευρωκοινοβούλιο συμπλήρωσε κάτι ψηλά με κάτι χάρη στι προτεραιότητε που πετύχαμε μέσω των πιστώσεων υποχρεώσεων και πράγμα το οποίο θα ενισχύσει το πρόβλημα των ε, Ρέστα Λικιντέ, ε, των ε, ΡΑΛ. Έχουμε όμως ε, προβλήματα για το 2012. Καταρχήν μπαίνουν σε ανταγωνισμό διάφορα προγράμματα ε, λόγω της αναζήτησης πόρων και έτσι δεν έχουμε μπορέσει να φτιάξουμε τους κατάλληλες, ε, να προετοιμαστούμε μάλλον καταλήλως για να βγούμε από την κρίση, για όταν θα βγούμε από την κρίση και επίσης δεν έχουμε κατάλληλα κονδύλια για να αναπτύξουμε διαρθωτικές προτεραιότητες. Επίσης για την εποπτεία ή για ένα πραγματικό σύστημα αντιμετώπισης της κρίσης, όλα αυτά αγνοήθηκαν τα παντελώς στον προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη επιβάλλουν τη λιτότητα στην Ένωση, όπως την επέβαλαν και στους πολίτες τους. Και οι σημερινές διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό είναι απλά το προήμιο για τα όσα θα συμβούν με, τον, ε, με το πολιετές πλαίσιο. Η κρίση εμπιστοσύνη με την αμφισβήτηση του Συμβουλίου των ε, νούμερων ε, που πρότεινε η Κομισιόν, πράγμα που σίγουρα θα σας ικανοποιήσει κύριε Επίτροπε, η η στάση αντίθετη με τις αρχές ε, ε, του προϋπολογισμού και με εμά είναι ε, προφανής για την κατάσταση που θα ακολουθήσει. Ωστόσο, ήδη οι πόροι νομίζω πως θα ήταν μια καλή λύση. Ανάμεσα στους καθαρούς συμβάλλοντες και στους υπολείπους υπάρχει σαφή διαφορά. Ο κύριος Μαρνέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρέπει με κάθε τίμημα να ευχαριστήσουμε τους εισηγητές που χρειάστηκε να διαπραγματευτούν χωρίς καμία πραγματική δυνατότητα, κανένα περιθώριο ελιγμού και παρόλα αυτά κατάφεραν να ολοκληρώσουν ένα τεράστιο έργο για να πετύχουν τους στόχους που είχε ορίσει το Ευρωκοινοβούλιο. Επιπλέον θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονό ότι υπάρχει ο προπολογισμό. Έχουμε προπολογισμό. Διανύουμε μια περίοδο κρίση και θα ήταν πραγματικά αντιπαραγωγικό το να είχαμε επιπλέον και μια δημοσιονομική κρίση. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στη σοφία του Κοινοβουλίου. Θα μπορούσαμε να έχουμε μπλοκάρει τα πάντα, αλλά δυστυχώς το Συμβούλιο δεν επέδειξε την ίδια σοφία. Σεβαστήκαμε τη συνθήκη της Λισαβόνας κατά τη διάρκεια αυτής της δημοσιονομικής διαδικασίας. Κάθε φορά όμως το ίδιο γίνεται το Συμβούλιο επιβάλλει τα νούμερα που θέλει για τις πιστώσεις πληρωμών και δεν μετακινείται από εκεί. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν νομίζω πως αυτός ο τρόπος να υπαγορεύει τα νούμερα και έπειτα να κατανέμει ανάμεσα στους διάφορους ε, πολιτικούς ευρωπαϊκούς τομείς είναι η κανονική φυσιολογική διαδικασία. Το κανονικό θα ήταν να αξιολογηθούν οι ανάγκες και έπειτα στη συνέχεια να υπολογιστεί προπολογισμό. Σίγουρα το Συμβούλιο έκανε μια δήλωση μέσω της οποίας δεσμεύεται να δεχτεί το διορθωτικό, με διορθωτικές επιστολές τη στιγμή όπου θα χρειαστούν τα χρήματα που δεν θα είναι διαθέσιμα μάλλον χρήματα για την εκτέλεση του προεκλογισμού όμως το Συμβούλιο δεν κράτησε το λόγο του αρκεί να δει κανείς τι έκανε το Συμβούλιο με τον διορθωτικό προπολογισμό 6 ε, και όταν ήρθε αυτός στο τραπέζι της συζήτησης. Δεν μπορούμε όμως να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατόν επίσης να μην εμπιστευόμαστε τα νούμερα που παρουσιάζει η Κομισιόν. Του χρόνου έχουμε δύο πολύ σημαντικές δημοσιονομικές διαδικασίες. Ε, τον προπολογισμό του 2013 και έπειτα το πολιετές ε, πλαίσιο. αν ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία θα είναι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριε Μαρινέσκου. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο, η κυρία, ο κύριος Σαμπάτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν πρέπει να υπογραμμίσουμε πως αυτή η συμφωνία για πρώτη φορά υιοθετήθηκε σε συμμόρφωση με τη νέα δημοσιονομική διαδικασία που ορίζει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ωστόσο για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε την ανάγνωση του Συμβουλίου για τις πληρωμές κάτω 2% φέτος, δηλαδή λιγότερο από το 2011 σε πραγματικούς όρους. Και είπαμε ότι αυτή η απόφαση είναι αντίθετη με την της με την πρόταση της Κομισιόν που κατέδειξε τις ανάγκες για το 2011. Ωστό, βέβαια, πετύχαμε τις πιστώσεις υποχρεώσεων που επιθυμούσαμε σε όλους τους τομείς σχεδόν. Ωστόσο, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο, κανονι... ο προϋπολογισμός στη διάρκεια της εκτέλεσής του. Είναι μια μέθοδος που δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χαράξει μεγάλους προσανατολισμούς, κυρίως στην έρευνα. Ε, να θυμίσω ότι ο κοινοτικό προπολογισμό παραμένει ένα μοχλό και παρά την πολιτική λιτότητα που ακολουθείται αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη και την οποία κατανοούμε, θα πρέπει να αναλάβουμε ως ένα μίνιμουμ δεσμεύσεων με ένα 4% επιστροφή στου πολίτε, ο ευρωπαϊκό προπολογισμό να μην αποτελεί μια μαύρη τρύπα, αλλά ένα εργαλείο κατανομή που επιτρέπει τι επενδύσει για το μέλλον. Σα ευχαριστούμε κυρία Μπάτ. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Καρβάλιο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι για την ε, συμφωνία που εξευρέθη στη συνδιαλλαγή και που το Συμβούλιο δέχτηκε για τον προπολογισμό του 2012. Ωστόσο, παραμένει το γεγονός ότι το Συμβούλιο συμφώνησε με το Κοινοβούλιο για 200 εκατομμύρια ευρώ από το μέσο ευελιξίας. Η χρήση αυτών των 200 εκατομμυρίων ευρώ ανταποκρίνεται στην, ε, ε, στο αίτημα του Κοινοβουλίου να τροφοδοτηθεί ανταγωνιστικότητα. Ανάμεσα στις διάφορες προτεραιότητες για το 2012 θα ήθελα να αναφέρω κάποια παραδείγματα όπως το πρόγραμμα για την πρόθεση του τουρισμού, η έρευνα, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Εράσμος Mundus και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ. Και η έρευνα σχετικά με αυτές. κυρία Ματέρα για δύο λεπτά. Επίτροπε, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μου και να συγχαρώ τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην ομάδα συνδιαλλαγής με το Συμβούλιο για την περίπλοκη δουλειά που χρειάστηκε να λυθεί υπόψη περίοδο, την περίοδο λιτότητας και τις δυσκολίες των προϋπολογισμών των κρατών μελών που ήδη δοκιμάζονται σκληρά. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης μπορεί να θεωρηθεί θετικό όσον αφορά τις προτεραιότητες της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ, όπως αυτό τις είχε προκαθορίσει. Κυρίως αναφέρομαι στην κατηγορία 1α που είναι ε, κατηγορία κλειδί για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και για την στήριξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου όπου η συμφωνία για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για το Life Learning και το Erasmus Mundus διατηρήθηκαν. Δεν μπορώ ωστόσο να δεχτώ ότι για το δεύτερο, δεύτερη διαδοχική χρονιά το Συμβούλιο έχει επιβάλει οριζόντιες περικοπές αμετάκλητες ε, κιόλας για όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού. 1,86% είναι η μείωση της, ε, των πληρωμών σε σχέση με το 2011 και αυτό είναι αντίθετο με τη γραμμή που προτείνει η Κομισιόν και που στόχο έχει την ε, οικονομική ανάκαμψη και που, την οποία στηρίζει έντονα αυτό το Κοινοβούλιο. Το να βασιστούμε στις προτεραιότητες σε μια στιγμή λιτότητας αντιπροσωπεύει σίγουρα μια νικηφόρο στρατηγική. Αυτό που διαφαίνεται ωστόσο από τη συνδιαλλαγή είναι μια ανισότητα ανησυχητική ανάμεσα τις ανηλυμένες υποχρεώσεις και τις, τα κονδύλια που όντως έχουν εγκριθεί. Το αποτέλεσμα αυτό κινδυνεύει να ε, δυναμητήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη για τη δυνατότητα να βρούμε ε, αλόβετη από αυτή την φάση μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών ε, δυσκολιών. Σας ευχαριστώ και τώρα έχει το λόγο για δύο λεπτά ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμε, κύριε Επίτροπε, κύριε Λεβαντόφσκι, συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση του προεπλογισμού αυτού. Γιατί πιστεύω ότι και για τα κράτη-μέλη μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα προ μίμηση. Για τι πληρωμέ θα πρέπει να συγκρινόμαστε με το μέσο όρο των πληρωμών στα κράτη-μέλη και με την ανάληψη υποχρεώσεων. ίσω θα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να ε, μην υπερβούν και εκείνα αυτή την οροφή που έχουμε επιβάλει και στους εαυτούς μας. Νομίζω λοιπόν από την αρχή τη διαπραγματευτική θα πρέπει να υπάρξει και ένας αυτοματισμός και ένας αυτοπεριορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να μην υπερχρεωνόμαστε και αυτόν τον αυτοπεριορισμό και την αυτοδέσμευση ε, να κληθούν και τα κράτη-μέλη να την αναλάβουν εθελοντικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι ε, το πρόγραμμα Έρασμος για τους δημοσιογράφους που το είχαμε εισαγάγει πέρυσι ως προπαρασκευαστική δράση. Χαίρομαι που το ε, υιοθέτησε η κυρία Κρούς και το πρόγραμμα αυτό για τους δημοσιογράφους αυτό το θέμα ανταλλαγής μεταξύ των ε, δημοσιογράφων από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα για να ενημερώνονται πώς ασκείται ευρωπαϊκή πολιτική στα διάφορα κράτη-μέλη και πώς προβάλλεται στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες, στα κοινωνικά δίκτυα. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να φέρουμε πιο κοντά τους δημοσιογράφους στην ε, πραγματική Ευρώπη. Χαίρομαι και για το πρόγραμμα Έρασμος ε, για νέους επιχειρηματίες γιατί εδώ δημιουργείται απασχόληση, νέες θέσεις απασχόλησης. Ε, δίκτυα καινούρια, κανεί γνωρίζει τους πελάτες του, τους προμητευτές Χαίρομαι επίσης ε, και για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ολυμπιάδα των νέων στο Ίνσμπρουκ. Είναι πολύ καλό να φέρνουμε κοντά τους νέους πέρα από σύνορα, ειδικά στον αθλητισμό που καλούνται να έχουν και κάποιες επιδόσεις. Όλα αυτά είναι σημαντικά για μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρουμπίκ. Για δύο λεπτά ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ε, ήλθε αυτή η συμφωνία κύριε Πρόεδρε, τη χαιρετίζω ιδιαίτερα λόγω της ε, οικονομικής ε, ύφεσης και κάμψης είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε αυτές τις ε, ρυθμίσεις. Ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορέσει να επιτευχθεί κάποια αύξηση του προϋπολογισμού. Θα ήθελα εγώ να εστιάσω την προσοχή μου στον αθλητισμό εδώ. Οι νέε γραμμές του προϋπολογισμού και επίσης για τα θαλάσσια θέματα Αυτά τα, οι νέες προτάσεις της κυρίας Δαμανάκη για τα θαλάσσια θέματα μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε νέες θέσεις εργασίας. Και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την ανάπτυξη ανανεώσιμων ενεργειών στον Ατλαντικό με την χρήση της αιωλικής ενέργειας και επίσης ενέργειας των κυμάτων. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με νέα υλικά και οι υπεράκτιες αιωλικές εγκαταστάσεις είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που υπάρχουν και επίσης να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε βιώσιμη αλληλεία που προέρχεται από τα δικά μας ύδατα και όχι να έρχεται από αμφισβητήσιμες πηγές. Για τον αθλητισμό θέλω να επικροτήσω αυτά που είπε ο κύριος ε, Ρούμπικ. Θα ήθελα να υπάρχει ένας έρασμος για τον αθλητισμό. Πρέπει να δώσουμε αρκετή σημασία, αρκετή με περισσότερη σημασία στη ικανότητα του αθλητισμού να ξεπερνάει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, ιδίω τις δυσκολίες σε επίπεδο υγείας. Όλοι ζητούν περισσότερα χρήματα για να κάνουν έρευνα και να θεραπεύσουν διάφορες ασθένειες. Η λύση είναι πολύ απλή. Η πρόληψη. Η πρόληψη ξεκινά με το να ζουν οι άνθρωποι με ένα υγιεινό τρόπο. Νους σώμα, τη γη. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Περνάμε στην διαδικασία Catch the Eye. Ε, Πρώτος ο κύριος Κοσλόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίρον και το Συμβούλιο και την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο εξευρέθη μια συμβαστική λύση για τον προπολογισμό του 2012. Προφανώ δεν έχουμε επιτύχει το επίπεδο το οποίο αρχικά είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παρόλα αυτά ήταν ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Θέλω επίση να συγχαρώ την Πολωνική Προεδρία γιατί συμμετέσχει και αυτή στις επιτυχίες αυτές διαπραγματεύσεις και προσπάθησε να μεσολαβήσει μεταξύ των θέσεων των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των θέσεων των κρατών μελών. Οι περικοπές λοιπόν δεν θίγουν την πολιτική συνοχής που είναι η πιο αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε καιρό κρίσης μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει επαρκές επίπεδο επενδύσεων. Με ένα τέτοιο προϋπολογισμό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε αποθεματικά και περιθώρια όπου δεν υπάρχει πλήρης εκταμίευσης και να έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε όλη τη δυνατότητα μέτρων για την απασχόληση. Ευχαριστώ. Κύριε Σουίξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με πολλά σχόλια σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012. Πιστεύω λοιπόν ότι οι προτάσεις του Συμβουλίου για τις πιστώσεις πληρωμών και απασχολήσεων και υποχρεώσεων ξεπερνούν τα εσκαμένα. Αν δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με την διοίκηση, τα πράγματα δεν είναι καθόλου θετικά. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την πρόταση του Συμβουλίου για τις ε, θέσεις που έχουν να κάνουν με τα αποθεματικά. Θα πρέπει να είναι επαρκή τα αποθεματικά. Και αυτό αφορά κυρίως τις κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την εξωτερική δράση. Ευχαριστώ. Ο κ. Μοργκάντη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω πω ο συμβιβασμό που επετεύχθη στη συνδιαλλαγή είναι αρκετά ικανοποιητικό. Αυξήθηκαν τα κονδύλια για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυξήθηκε επίση και το κονδύλι για το Frontex, την υπηρεσία ελέγχου για τα ευρωπαϊκά σύνορα. Σε μια περίοδο αντικειμενικών δυσκολιών δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε περισσότερο και θα έλεγα μάλιστα ότι θα ήταν ε, καλύτερο να καταργηθούν και κάποιε δαπάνε που δεν θεωρώ ότι είναι Όπω όπως ας πούμε η αύξηση της αναπτυξιακής συνεργασία με την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, είναι σκανδαλώδη η περαιτέρω αύξηση των ε, κονδυλίων για τη στήριξη τη τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να νομιμοποιεί έναν λαό ο οποίος παράνομα κατέχει εδάφη τα οποία δεν του ανήκουν. Εν πάση περιπτώσει δεν, έγινε, δεν είναι μεγάλη η δαπάνη για τα κράτη-μέλη που δοκιμάζονται ε, σκληρά από την κρίση και αυτό ήταν το πιο σημαντικό που έπρεπε να επιτύχουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Μοργκάντη. Ναι, κύριε Ρούμπιγκ. Διαδικαστικό έχετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα μόνο να σας ανακοινώσω ότι μου κλέψαν τα ακουστικά μου από το έδρανό μου. Δεν είναι δυνατόν σε αυτό το κοινοβούλιο συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Ήταν δικά μου, ιδιωτικά, τα προσωπικά μου ακουστικά εξαφανίστηκαν. Να δούμε, θα το λύσουμε κύριε Ρούμπιχ. Θα ενημερώσουμε την ασφάλεια. Αλλά πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικά αυτά τα πράγματα. Το λόγο έχει ο Επίτροπος κύριος Λεβαντόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Συζητούμε ένα πολύ μετριοπαθή ε, ε, προπολογισμό συγκρατημένο για το 2012 κάτω του 1% ε, του ΑΕΠ των κρατών μελών, παρόλο που έχουν αυξηθεί και οι αρμοδιότητες από τις συνθήκες Λισαβόνας και οι προκλήσεις που αξίζει να έχουν κοινή απάντηση. Ονομαστικά μπορεί να αυξάνεται ο προπολογισμό, αλλά σε πραγματικούς όρους μειώνεται. Δεν ζητούμε ούτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε για το Κοινοβούλιο επιπλέον. Αρχίζουμε οικονομίες. 94% ε, ζητούμε για επιχειρησιακές ε, δράσεις, πολύ διαφορετικής φύσεως από ότι οι κρατικοί προϋπολογισμοί. Και θέλω να απαντήσω σε ορισμένους ομιλητές ότι μας στυλιτεύουν και μας κατηγορούν ότι αυξάνουμε τον προπολογισμό ενώ οι χώρες εξοικονομούν. Αυτό δεν ισχύει γι' αυτό. Για τέσσερις χώρες, ε, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτοκαλία και Ιρλανδία, οι άλλοι ε, προπολογισμοί των κρατών μελών αυξάνονται συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και των κάτω χωρών διότι παρόλες τις οικονομίες έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις σε αιτήσια βάση να καλύπτουμε και στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό ισχύει πάγια με τη μεγάλη διαφορά ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός είναι πάντα ισοσκελισμένος και δεν μπορεί να φορτώνεται την κακή δημοσιονομική διαχείριση των κρατών μελών και ε, γίνονται και επενδύσεις, όπως πολύ καλά εξήγησε ε, η κυρία Γένσεν ή ο κύριος Βόν από την Ουαλία. Δεν πούμε που το επαναλαμβάνω τόσο συχνά, αλλά από ό,τι φαίνεται ορισμένα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν τη συνήθεια να ε, κάνουν ε, την κριτική τους και να φεύγουν πριν ε, πάρουν τις απαντήσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε Από το Συμβούλιο το λόγο τώρα έχει ο κύριος Δομινίκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση για τις πιστώσεις πληρωμών μπορεί να γίνεται και πάντα θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι δεν θα είναι ικανοποιημένοι. Και το ίδιο ισχύει και για τους ίδιους τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Κάποιοι θα είναι πάντα γκρινιάριδες θα διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ορισμένα θέματα δεν έχουν καλυφθεί με επαρκή κονδύλια. Σας πεθυμίζω όμως ότι έχουμε μια διαφορετική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Για όλη αυτή τη διαδικασία του προπολογισμού για το 2012 υπάρχουν δύο σημαντικά μηνύματα τα οποία μπορούμε να εξαγάγουμε. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα τονίσω τώρα και αξίζει να τα θυμάστε κι εσείς. Καταρχήν, στην φετινή διαδικασία του προϋπολογισμού επιβεβαιώσαμε ότι μπορούμε ακόμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλύουμε δύσκολα προβλήματα. Χρησιμοποιώντας την κοινοτική ή ενωσιακή μέθοδο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό λοιπόν μήνυμα γιατί ακολουθήσαμε πιστά αυτά τα οποία προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας για να επιτευχθεί η συμφωνία. Δεν χρειάστηκε καμία περαιτέρω δράση που να ξεφεύγει από τον περίγυρο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις τωρινές <clears throat> συγκυρίες αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να το εξάρουμε και το καταδείξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι λειτουργεί ακόμα η κοινοτική, η ενωσιακή μέθοδος. Κάτι ακόμα, το γεγονός ότι παρά τις επικρίσεις που έχουν ακουστεί για τον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 6, είναι σαφές ότι οι υποχρεώσεις που έχουν συναυθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, οι δεσμεύσεις αυτές πράγματι τήρούνται. Μπορεί κανείς να μην συμφωνεί για τα 200 εκατομμύρια, για το συγκεκριμένο αριθμητικό ποσό. Όσοι όμως έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία συνδιαλλαγής, θυμούνται ότι αυτό ήταν ακριβώς το ποσό για το οποίο συζητήσαμε. Αν λοιπόν τη στιγμή που παίρνουμε αποφάσεις. Μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτά τα ποσά χρειάζεται ο προπολογισμό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν το αντικείμενο λοιπόν της συζήτησης, όχι αν θα έπρεπε να δώσουμε χρήματα, αλλά πόσα χρήματα θα έπρεπε να δώσουμε. Κατά τη δική μου λοιπόν κρίση, αυτά τα δύο σημεία που ανέφερα είναι πολύ σημαντικά συστατικά της διαδικασίας και πρέπει να τα θυμόμαστε. Είμαστε τώρα επιτυχείς στο να εφαρμόσουμε τις διατάξεις της ε, συνθήκης Λισαβόνας και αυτό θα πρέπει να το χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Ντομινίκ. Ο κύριος Λαμασίρ έχει το λόγο. Για να έχετε τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου στην ανάλυση του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη των 27 είναι η χρήσιμη Ευρώπη και η Ευρώπη που λειτουργεί ακούμε εδώ και εκεί να εκφράζονται διάφορες επιθυμίες να συγκεντρωθούν ορισμένα κράτη-μέλη για να προχωρήσουν ε, λειτουργώντας και εργαζόμενα ε, λίγα μέλη σε κάποιους τομείς. Η Ευρώπη όμως που λειτουργεί σήμερα είναι Ευρώπη των 27 και σε αυτό το κρίσιμο τομέα βρήκαμε συμφωνία, καταλήξαμε για να έχει προπολογισμό η Ένωση για το 2012, αυτή είναι καλή είδηση και Κατά τα λοιπά, θυμίζω, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το σχέδιο προπολογισμού και το συγχαίρω. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει εντό ολίγων λεπτών. Είναι τρει οι διαδοχικέ ψηφοφορίε. Μία για την προσαρμογή τη Διοργανική Συμφωνία, μία για τον προπολογισμό αυτό καθ' αυτό του 2012 και μία ψηφοφορία για το διορθωτικό προπολογισμό για το 2011 και οι τρεις αυτές ψηφοφορίες είναι τμήμα μιας πολιτικής συμφωνίας. Και καλώ τους συναδέλφους με μεγάλη πλειοψηφία να υποστηρίξει, που βεβαίως δεν θα αγγίξει την ομοφωνία του Συμβουλίου, αλλά μπορεί να την προσεγγίσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαμασούρ μου. Ολοκληρώνει τη συζήτηση εδώ για τον προπολογισμό. Διάλειμμα 5 λεπτών και στις 12 ακριβώς αρχίζουν οι ψηφοφορίες.